Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Λίγοι είμαστε στην αίθουσα, αλλά νομίζω ότι είμαστε αρκετοί παρόντες για να ξεκινήσουμε. Και αρχίζουμε με το σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης, την έγκρισή της. Δεν υπάρχει καμία τήρηση. Φαντάζομαι πάμε στο σημείο 2 που είναι οι ανακοινώσει του Προέδρου. Λοιπόν, έχουμε και το web streaming, web streaming συγγνώμη, δηλαδή θα μεταδίδεται όλη η συνεδρίασή μας. Είναι η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας πριν από τις εκλογές. Όλα τα μέλη είναι προσκεκλημένα στο 3 σε 050 όλοι, όλα τα μέλη και όλοι οι αναπληρωτές εδώ όταν τελειώσει, τελειώσουν οι, συνεδρι, οι συνεδριάσεις μας. Θα πιούμε ένα ποτό και μετά στις 6.30 όλα τα μέλη επίσης τα προσκαλούμε, τα προσκαλώ εγώ ε, στο, στην τραπεζαρία των μελών, τα μέλη και οι αναπληρωτές. Τώρα πάμε στο σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων που έλαβαν χώρα από τις 23 ε, έως τις 25 Ιουνίου 2008, 21 και 22 Ιανουαρίου 2009, 9 με 11 Φεβρουαρίου 2009, 16 Φεβρουαρίου 2009 και 16 Μαρτίου 2009 θεωρούμε ότι έχουν εγκριθεί εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις που θα εκφραστούν μέχρι το τέλος της παρούσας συνεδρίασης. Και τα πρακτικά της σημερινής μας συνεδρίασης, της σημερινής και της αυριανής δηλαδή, θα προωθηθούν σε όλα τα μέλη έτσι ώστε να εγκριθούν μέσα στα πλαίσια μιας γραπτής διαδικασίας. Τώρα πάμε στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης πρότυπα ποιοτητα και ασφάλεια των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτηση, δίδοντας το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Φρίντα Μπριπόους, που έχει και το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα γιατί προσθέθηκε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη και έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε την ανταλλαγή απόψε. Είναι γεγονός ότι δεν είναι πολυπληθής η προσέλευση στην συνεδρίασή μας, αλλά είναι εκλεκτοί οι συνάδελφοι και νομίζουμε, νομίζω ότι μπορούμε να διεξέλθουμε το θέμα αυτό. Οι δεωρές οργάνων και οι μεταμοσχεύσεις, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει μια μακρά ιστορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 10 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε βρισκόταν στα πλαίσια της ε, συνθήκης του Μάστριχτ και είχε ήδη θεσπίσει μια σειρά από μέτρα για την ποιότητα των ιστών και των οργάνων που είχαν να κάνουν με τις μεταμοσχεύσεις και επίσης για την αιμοδοσία και την ε, παροχή ιστών έχουν επέλθει σημαντικές πρόοδοι σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις. Το 2003 και 2004 έχουν εγκριθεί μια σειρά από οδηγίες. Και για τα όργανα έχει αποφασιστεί να ακολουθήσει μια διαφορετική οδό η Κομισιόν η οποία ίσως να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να καλυφθούν οι δωρεές και μεταμοσχεύσεις οργάνων, που φυσικά εδώ είναι πιο δύσκολο το ζήτημα αυτό, πιο πολύπλοκο, διότι έχουμε διαφορετικές προδιαγραφές οι οποίες ισχύουν στα κράτη-μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη δική του πλευρά και ιδίω ορισμένα μέλη της Επιτροπής καταναλωτών και δημόσιας υγείας έχουν ζητήσει κάτι επανάληψη από την Κομισιόν να επεξεργαστεί προτάσεις βάσει των οποίων θα μπορούσαν να προκύψουν κοινέ ρυθμίσεις οι οποίες θα μπορούσαν να διέπουν μια καλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό μπορώ να διαπιστώσω με μεγάλη ικανοποίηση το ότι η Κομισιόν έχει αναφέρει ότι θα παρουσιάσει ως Νούπο μια ανακοίνωση για τα θέματα αυτά, καταρχήν για να υπάρξει ένα σχέδιο δράση για την βελτίωση της ασφάλειας των ε, μεταμοσχεύσεων και δωρεών οργάνων, ώστε να υπάρξει καταρχήν μια ανταλλαγή απόψεων και πελσίστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και επίσης να υπάρξουν και τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδιστεί το εμπόριο, το λαθρεμπόριο καλύτερα, οργάνων. Αυτά είναι θέματα λοιπόν τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε στην Επιτροπή μας έχουμε το ψήφισμα του 2008 ήδη από την Επιτροπή μας που ήταν εισηγητής τότε για το ίδιο θέμα ο κύριος Σαδάμου. Και υπάρχει ένα οδηγό νήμα το οποίο δημιουργείται βάσει αυτής της ε, πρότασης, αυτής της ε, ε για να μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερες δωρεά, οργάνων στην Ευρώπη, γιατί τα όργανα αυτά τα οποία δίνονται από τους δότες σώζουν πολλές ζωές στην Ευρώπη. Δυστυχώς υπάρχει μια έλλειψη δοτών και είναι πάρα πολλοί Ευρωπαίοι οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους αναμένοντας να βρουν δότες οργάνων. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε εδώ ότι η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο για να καλυφθεί το πρόβλημα αυτό. Τον προηγούμενο Δεκέμβρη η Κομισιόν δημοσίευσε μια πρόταση ώστε να υπάρξει μια οδηγία εν καιρό και ένα σχέδιο δράσης και στις 3 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα προτού δημοσιευτεί αυτό, αυτή η ανακοίνωση της Κομισιόν είχαμε συγκεκριμένη πληροφόρηση για το θέμα αυτό από τον αρμόδιο επίτροπο σε ένα δείπνο εδώ στο Κοινοβούλιο. Χαίρομαι λοιπόν που γνωρίζω πλέον ότι η Κομισιόν φαίνεται ότι έχει συμπεριλάβει στην έκθεσή της πολλές από τις απόψεις που είχε διατυπώσει τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο τέλος Δεκεμβρίου εγώ ανέλαβα την εισηγεσία αυτού του θέματος και αυτό μου έδωσε μια περαιτέρω ευκαιρία να συζητήσω τα θέματα που διαλαμβάνει η πρόταση της Κομισιόν με διάφορους εμπλεκομένους ε, δημοσίες αρχές, ιατρούς, εκπρόσωπους επαγγελματικών κλάδων, ε, φαρμακευτικών εταιριών κτλ. Και σε γενική γραμμή μπορώ να πω ότι η αντίδραση όλων αυτών των φορέων ήταν ιδιαίτερα θετική. Αυτό το οποίο πρέπει να πράξουμε τώρα είναι να ελέγξουμε αυτές τις προτάσεις με πιο ενδελεχή τρόπο, να διευκρινίσουμε τα σημεία που αυτό είναι απαραίτητο και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και την πρόταση αυτή όπου αυτό απαιτείται. Θα ήθελα να τονίσω επίσης κύριε Πρόεδρε ότι είναι λυπηρό και ελπίζω ότι συμφωνούν και οι συναδελφοί μου ότι δεν έχουμε επαρκή χρόνο για να μπορέσουμε να περατώσουμε τη διαδικασία λήψη απόφασης για το νομοθέτημα αυτό πριν από τις εκλογές. Υπάρχει ένα συζητητής από τη δική μας πλευρά για αυτή την οδηγία, αλλά όχι για το σχέδιο δράσης. Αυτό είναι κρίμα λοιπόν. θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό από την επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Αλλά πρόκειται για δύο θέματα τα οποία είναι αλληλένδετα σε σχέση με το περιεχόμενό τους και είναι κρίμα που δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε από κοινού. Τι να κάνουμε όμως. Αυτό είναι λοιπόν το πλαίσιο μέσα στο οποίο η απόφασή μας ήταν να μην υποβάλουμε ένα σχέδιο έκθεσης από τη δική μας πλευρά, απλώς να κάνουμε μια συζήτηση για να διαφανούν οι γενικές κατευθύνσεις στην Επιτροπή μας και έχω συντάξει και ένα έγγραφο εργασίας με αυτό το σκοπό που ελπίζω θα μπορέσει να ευνοήσει την επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας. Ελπίζω ότι όλοι είχαν τον καιρό να το διαβάσουν. Έχει μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Δεν πρόκειται να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτού του εγγραφού. Αλλά θέλω να τονίσω ότι πρώτα στις Κομισιόν ακολουθεί μια ευρεία προσέγγιση και αυτό το οποίο εμένα προς τα πλαίσια της Επιτροπής μας είναι να υπάρξουν οι μηχανισμοί οποίοι θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια των οργάνων σε όλα τα κράτη-μέλη και θα μπορέσουν παρόλα οι αρμόδιες αρχές στα κράτη-μέλη να έχουν επαρκές περιθώριο για να εφαρμόσουν στις συγκεκριμένες συνθήκες της κάθε χώρας τους κανόνες αυτούς. Υπάρχουν ορισμένα σημεία στα οποία θα ήθελα να σταθώ και να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό. Είναι ζητήματα στα οποία μπορεί να απαιτείται περαιτέρω διευκρίνηση ή περαιτέρω συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ευελιξία μέσα στο ψήφισμα το οποίο θα προέλθει από εμά. Να τονιστεί η ανάγκη ευελιξίας γιατί αυτό είναι απαραίτητα να υπάρχει μέσα στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ορισμένα τμήματα της πρότασης της Κομισιόν, παραδείγματος χάρη τεχνικά προγράμματα εξασφάλισης ποιότητος, καθώς και τα παρατήματα είναι ιδιαίτερα λεπτομεριακά. Χαίρομαι για το γεγονός ότι τα παρατήματα δεν θα αντιμετωπιστούν με τη διαδικασία της επιτροπολογίας, μπορούν να τύχουν αλλαγών τα παρατήματα μεταγενέστερα, εάν αυτό είναι απαραίτητο στο φως των προόδων της ιατρικής επιστήμης. Αυτή τη στιγμή τα παρατήματα περιλαμβάνουν όλο τον κατάλογο προϊόντων και όλες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες ώστε να δώσουν τα απαραίτητα εργαλεία στους γιατρούς ώστε να αποφασίσουν κατά πόσον ένα όργανο μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο ή όχι. Ξέρω ότι ορισμένοι μπορεί να έχουν κάποιες ανησυχίες για τα θέματα αυτά. Ξέρω ότι ορισμένοι θεωρούν ότι όλα αυτά αποτελούν υπερβολική γραφειοκρατία. Ίσως εδώ η Κομισιόν μπορεί να μας δώσει τη δική της ε, άποψη για τα ζητήματα αυτά. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο για μένα ήταν πολύ σημαντικό στην πρόταση αυτή είναι η σχέση μεταξύ των εθνικών αρχών και του Ευρωπαϊκού Φορέα για την ανταλλαγή ε, πληροφοριών στα θέματα αυτά. Νομίζω ότι οι εξουσίες που δίνονται στις εθνικές αρχές είναι ιδιαίτερα φιλόδοξες. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοιου είδους αρχές στα περισσότερα και γι' αυτό είναι απαραίτητο να εξετάσουμε κατά πόσο οι ανταλλαγές μεταξύ τωρινών, ε, ανταλλαγές οργάνων μάλλον, μεταξύ εθνικών αρχών και ευρωπαϊκών τραπεζών οργάνων μπορούν να λάβουν χώρα. Ένα τρίτο σημείο είναι το θέμα της σύνδεσης αυτής της ε, πρότασης με άλλα νομοθετήματα. Νομίζω ότι λάβουμε υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των μεταμοσχεύσεων και το ευαίσθητο του συστήματος το οποίο διέπει τις μεταμοσχεύσεις οργάνων και τους καταλόγους για τα όργανα, ίσως θα έπρεπε να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα προβλέπει εξαιρέσεις μέσα στην οδηγία αυτή που επεξεργάζεται ο συζητητής, ο συνάδελφός μου κ. Μπόης, για την ε, ε, μεταμόσχευση οργάνων στα πλαίσια της διαμεθοριακής παροχής ιατρικών φροντίδων και θεραπείων. Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο και στο θέμα το οποίο συζητούμε σήμερα. Επομένως θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα των εξαιρέσεων και επίσης είναι σημαντικό να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε σαφώς την εμβέλεια αυτής της οδηγίας γιατί ορισμένοι έχουν την τάση να ερμηνεύουν αυτό το νομοθέτημα με ιδιαίτερα περισταλτικό τρόπο. Εγώ έχω θέσει το ερώτημα του γιατί η κατανομή των οργάνων στους ε, ασθενείς εκφεύγει της ε, σφαίρας εφαρμογής αυτής της ε, έκθεσης και γιατί δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη το θέμα της των αποτελεσμάτων που μπορούν να προκύψουν από μια μεταμόσχευση. Υπάρχει επίσης και μία αναφορά σε, στα δίκτυα τα οποία συνδέουν τις ε, εθνικές αρχές για να υπάρξει μεταλαμβάνευση βελτίστων πρακτικών. Για μένα αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να συζητήσουμε την ε, ανταλλαγή βελτίστων ιατρικών πρακτικών κατά τρόπον ώστε να επιτύχουμε τον βασικό στόχο αυτής της οδηγίας που είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των οργάνων για όλους τους ασθενείς της Ευρω... στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης να κάνει περισσότερα όργανα διαθέσιμα. Και επίσης είναι απαραίτητο να ερευνηθούν και οι μέθοδοι για την πρόληψη της απόρριψης των μεταμοσχευμένων οργάνων. Νομίζω ότι και στο έγγραφο αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει επιπλέον το θέμα των ορισμών. Κάποιοι ορισμοί ίσως θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίες. Παραδείγματος χάρη, τι είναι ένα όργανο. Ο ορισμός του όργανου. Και το τι, πώς ακριβώς καθορίζεται τι είναι δότης και τι είναι όργανο. Ίσως θα θέλαμε να προσθέσουμε εδώ πέρα και μια καλύτερη διατύπωση λέγοντας παραδείγματος χάρη ότι το επίπεδο της εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα αυτό όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 θα πρέπει να διατυπωθεί καλύτερα και μετά υπάρχει η ενζωή ε, δωρεά οργάνων και στο άρθρο αυτό, το αρμόδιο του άρθρο 15, πρέπει να είμαστε λιγάκι σαφέστεροι. Αυτή Τη στιγμή το άρθρο, όπως είναι διατυπωμένο, λέει ότι μία δωρεά εν ζωή δεν πρέπει να την χάνει αντιτίμου. Δεν μπορεί να καταβάλλεται το αντίτιμο μια τέτοια δωρεά και πιστεύω ότι αυτό είναι σωστό. Αλλά στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρσι είχαμε τονίσει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες κάποιο αντιστάθμισμα, κάποια αποζημίωση μπορεί να καταβάλλεται και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η πληρωμή καταβάλλεται μονάχα ως αποζημίωση και καλύπτει μονάχα την ε, απόδοση των εξόδων στα οποία υποβάλλεται ο δωρητής και οποιαδήποτε ε, μειονεκτήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν από αυτή την ε, πράξη δωρεάς. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Ένα τελευταίο σημείο, τα μητρώα και η χνηλασιμότητα. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στη σημασία του να υπάρχουν τέτοια μητρώα, να υπάρχει ανιχνευσιμότητα για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο οργάνων. Θα μπορούσαμε να έχουμε λοιπόν ένα πανευρωπαϊκό σύστημα ταυτοποίησης οργάνων. Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει από τους οργανισμούς ανταλλαγής οργάνων. Θα μπορούσαν αυτοί να βοηθήσουν, να μας δώσουν κάποια περαιτέρω στοιχεία και προτάσεις για ένα τέτοιο ευρωπαϊκό σύστημα και αυτό ίσως μπορούμε να το συζητήσουμε και πάλι στα πλαίσια της συζήτησης του σχεδίου δράσης. Εν κατακλείδη, κύριε Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω ορισμένε σκέψει. Προσωπικά νομίζω ότι η οδηγία και το σχέδιο δράση είναι ένα σημαντικό θετικό βήμα προ τα εμπρό. Μπορούν να μα βοηθήσουν να αυξήσουμε τον αριθμό των δυνητικών δόρυτων στην Ευρώπη, αλλά μέσα στα πλαίσια τη εξασφάλιση τη ασφάλεια στην Ευρώπη θεωρώ ότι όλο αυτό το θέμα παρόλα αυτά θα πρέπει να τεθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και είναι απαραίτητο επίσης να εξετάσουμε και τις αιτίες που οδηγούν σε μια ζήτηση οργάνων για μετανάστευση. Πρόσφατα είχαμε μιλήσει σε μια ομάδα εργασίας σε ό,τι αφορά την υγεία των νεφρών, όπου εγώ προείδρευα και μας είπαν ότι υπάρχουν περίπου 250.000 Ευρωπαίων που έχουν προβλήματα με τα νεφρά που μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με μεταμόσχευση, ούτε καν αιμοδιάλυση. Ένα 10% όλων των Ευρωπαίων έχουν κάποιο είδος χρόνιας νεφρίτιδος και αν δεν μπορούμε να εντοπίσουμε αυτές τις ασθένειες και να τις αντιμετωπίσουμε θεραπευτικά, μερικοί από αυτούς τους ανθρώπους εν καιρό θα χρειαστούν μεταμόσχευση νεφρών. Πρέπει να υπογραμμίσουμε λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει συνειδητοποίηση και πρόληψη για την ε, αποτροπή τέτοιου είδους ασθενειών όπως είναι η νεφρική ανεπάρκεια αλλά επίσης και καρδιοαγγειακών ασθενειών και άλλων ασθενειών οι οποίες συνδέονται με την ανάγκη μεταμόσχευση. Θα ανακλείσω εδώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ για την προσοχή σας και με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσω τα σχόλια ή τις ερωτήσεις που μπορεί να έχουν οι συναδελφοί μα και ελπίζω να είναι επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ. Thank you very much. ευχαριστώ πολύ. Συνήθως τώρα δίνω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές. Αλλά δεν βλέπω κανέναν να είναι παρόντα. Έχω άλλο ονόματα στον κατάλογο μου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την ανταλλαγή απόψεων με, δίνοντας το λόγο στην κυρία Πατρίτσια Κόκο από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ της Κομισιόν. Κυρία μου, έχετε το λόγο μέρος της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτή την πολύ επικοδομητική και υποστηρικτική ανάλυση της πρότασης της Κομισιόν για την ποιότητα και την ασφάλεια των οργάνων για μόσχευση. Τα βασικά σημεία έχουν πολύ σωστά φωτιστεί από την εισηγήτρια και χαιρόμαστε που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Ε, πρώτα απ' όλα σημείωσα ότι η συγγήτρια καλωσορίζει την ε, πρόταση. Επίσης, σημείωσα ότι θεωρεί ότι η πρόταση αφήνει αρκετή ευκαμψία όπως πρέπει στα κράτη-μέλη ώστε να εφαρμόσουν τις διατάξεις χωρίς να αναστατώσουν το εθνικό του σύστημα όταν αυτό ήδη υφίσταται. Σε σχέση με τις αποσαφηνίσεις που ζητήθηκαν θα προσπαθήσω να απαντήσω στα 7 σημεία που τέθηκαν. Το πρώτο σημείο αφορούσε την απαραίτητη ευελιξία. Λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα το γεγονός ότι ορισμένα σημεία ίσως αναπτύχθηκαν υπερβολικά με υπερβολική λεπτομέρεια, ειδικότερα δε ο κατάλογος των τεστ και τα εθνικά προγράμματα ποιότητας. Όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα ποιότητας, πιστεύουμε ότι πρέπει να υφίστανται. Δεν πρέπει να δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά πρέπει να δώσουμε κάποιες ενδείξεις σε σχέση με το τι προσδοκούμε, διότι όπως είπε η συγγήτρια, ένας από τους έμεσους και τονίζω το έμεσους φόρους, ε, του στόχους με συγχωρείτε, ε, διότι η νομική βάση δεν μας επιτρέπει να κάνουμε διαφορετικά, είναι να μειώσουμε το παράνομο ομπόριο οργάνων. Ένα λοιπόν από τα σημαντικά σημεία για την καταπολέμηση αυτή είναι να έχουμε συστήσεις, συστήματα τα οποία μπορούν να υπαλληθεύονται και να ελέγχονται. Έτσι κάνει κανείς τη δουλειά των ε, λαθρεμπόρων δύσκολη και αυτό είναι ακριβώς ο στόχος. Τώρα, ο χαρακτηρισμός των οργάνων που βρίσκονται στο παράρτημα. Αυτός βασίζεται στα συμπεράσματα ενός προγράμματος που εφάρμοσε η Κομισιόν με κάποιους εμπειρογνώμονες και αντανακλά τη σημερινή κατάσταση εξέλιξης και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Αυτά τα τεστ ήδη πραγματοποιούνται και αποτελούν το σύνολο των όσων είναι απαραίτητα να πραγματοποιηθούν για να γίνει αξιολόγηση του κινδύνου. Δεν ε, θέτουμε πρότυπα. Λέμε ότι όταν πρόκειται να κάνουμε αξιολόγηση του κινδύνου για το κατά πόσο ένα όργανο συγκεκριμένο είναι κατάλληλο για έναν ασθενή, αυτή πρέπει να είναι η βάση της αξιολόγηση. Τώρα, όσον αφορά τη σχέση μεταξύ αρμοδίων αρχών και οργανώσεων ε, οργάνων μεταμόσχευσης αναγνωρίζουμε την ύπαρξη και των αρμόδιων αρχών και των οργανισμών μεταμόσχευσης και δημιουργούμε και μια σύνδεση μεταξύ τους ώστε οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να εκχωρούν στους οργανισμούς μεταμόσχευσης κάποια από τα έργα ή τις ενέργειες σε σχέση με τη δωρεά οργάνων. Τώρα, γιατί το θέμα της διασυνοριακής κινητικότητας των ασθενών δεν εξετάστηκε εδώ. Εμείς στην πρότασή μας αναφερόμαστε στην ποιότητα και την ασφάλεια των αργώνων των οργάνων. Μπορεί συνεπώς να αναφέρεται και στην κινητικότητα των οργάνων, αλλά δεν έχει σχέση με την κινητικότητα των ίδιων των ασθενών. Ε, καλύπτεται αυτό από ένα άλλο πλαίσιο, το οποίο το γνωρίζετε άλλωστε πολύ καλά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, και αναφέρομαι στην τέταρτη ερώτησή σας, ε, σε ορισμένε περιπτώσεις θεωρείται ότι το εύρος είναι στενό και ότι η κατανομή των αργώνων έχει αποκλειστεί. Και εδώ είμαστε στη λεπτή γραμμή που χωρίζει το τι είναι απαραίτητο για τους ασθενείς και τι μπορεί να γίνει με αυτό το νομικό πλαίσιο και τι πρέπει να αφαιθεί στα χέρια των κρατών μελών. Πιστεύουμε ότι το σύστημα καταλωμής των οργάνων αφορά την επικουρικότητα και την εθνική οργάνωση του κάθε κράτου μέλους. Ακόμη είχατε μια ανησυχία για την απόρριψη οργάνων. Δεν κατάλαβα πολύ καλά ομολογώ. Ε, σας απασχολεί η απόρριψη των οργάνων ώστε να μην γίνει μεταμόσχευση ή η απόρριψη από τον ασθενή στον οποίο έχουν μεταμοσχευστεί. Η απόρριψη των οργάνων πριν από τη μεταμόσχευση βασίζεται στην αξιολόγηση του κινδύνου. Βεβαίω υπάρχουν τα φάρμακα τα οποία παρεμποδίζουν την απόρριψη και ε, βεβαίω υπάρχει και σχετική νομοθεσία που το διέπει. Έγινε και ένα σχόλιο σε σχέση με τους ορισμούς, ότι κάποιοι ορισμοί ενδεχομένω χρειάζονται βελτίωση. Προσπαθήσαμε να είμαστε συνεπείς μεταξύ των διαφόρων πλαισίων ε, και οι ορισμοί που περιλάβαμε σε αυτή την πρόταση είναι συμβατοί με τους ορισμούς στην οδηγία ιστών και κιτάρων και είναι σημαντικό ε, κείμενα τα οποία εγκρίνονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να είναι συμβατά μεταξύ τους. Ο χαρακτηρισμός των οργάνων θα μπορούσε να επικαιροποιηθεί με την επιτροπολογία και αυτό είναι σαφές με το άρθρο 25, γι' αυτό και δεν το επαναλαμβάνουμε για να απλουστεύσουμε το νομοθέτημα. Προσπαθούμε να αποφύγουμε επαναλήψεις ρυθμίσεων που ήδη ισχύουν. Είναι διατάξεις οι οποίες αναφέρονται ήδη αλλού για να, και δεν τις επαναλαμβάνουμε για να μην προκαλέσουμε σύγχυση. Στο, επίσης ε, στο έκτο σχόλιο σας αναφερθήκατε στην αποζημίωση των ζώντων δοτών η Κομισιόν σε σχέση με αυτό το θέμα θεώρησε ότι ε, δεν εμπίπτει στο πεδίο της ασφάλειας και της ποιότητας των οργώνων το να αναφερθούμε σε αυτό το ζήτημα. Περιελήφθη στο, στην οδηγία ιστών και κοιτάρων και το λαμβάνουμε υπόψη μας. Τώρα, όσον αφορά το λαθρεμπόριο, όπως σας είπα και στην αρχή, δεν μπορούμε να έχουμε άμεσο στόχο μέσω αυτής της πρότασης την καταπολέμηση του λατρεμπορίου, Αλλά έμεσα σίγουρα καθιστά πολύ δύσκολη τη ζωή για τους εμπόρους οργάνων. Είμαστε σίγουροι ότι θα συμβάλλει ή θα μειώσει πραγματικά στο ελάχιστο το παράνομο εμπόριο οργάνων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω ότι είναι εδώ ο βοηθό τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αποστασία των Δεδομένων, ο κύριο Χάστινγκ και ο κύριο Τζοβάνι Μπουταρέλη. Θα ήθελα να του ζητήσω να πάρει, το λόγο, εάν και εφόσον το επιθυμεί. Α. Thank you, Mr. Chairman. I would like to thank you. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια, διότι έδωσε στην υπηρεσία μας την δυνατότητα να προχωρήσει αυτή την ανταλλαγή απόψεων μετά τη γνωμοδότηση που είχαμε υιοθετήσει στις 5 Μαρτίου. Η, η ευρωπαϊκή αυτή υπηρεσία επίβλεψης και των προσωπικών δεδομένων είναι στη διάθεση σας για περαιτέρω συζητήσεις ασχολούμεθα με προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα που αφορούν ε, θανόντα και ζώντα άτομα, δεδομένα που πολλές φορές είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και ευάλωτα. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων γίνεται σε εθνικό επίπεδο στα κράτη-μέλη και αυτή ρυθμίζεται ήδη από την Εθνική Νομοθεσία που εφαρμόζει μια γενική οδηγία, την οδηγία 95-40-46. Και η πρόταση ε, αυτή αφορά για την, την προστασία των δεδομένων που αφορούν τους ε, δότες και τους λήπτες των οργάνων. Εμείς ε, υποστηρίζουμε τέτοιου είδου προτάσεις όμως θέλουμε να γίνουν κάποιες ε, αλλαγές. Έχουμε υποβάλει για αυτό το λόγο τροπολογίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων. Πιστεύουμε ότι οι προτάσεις πρέπει να είναι καλύτερα εναρμονισμένες και να λαμβάνουν υπόψη τον, τους στόχους, τους σκοπούς της πρωτοβουλίας αυτής. Συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει ανάγκη να επιτευχθεί ε, μια σωστή ισορροπία ανάμεσα σε μια επαρκώς ευέλικτη οδηγία, έτσι όπως αναφέρεται και στο κείμενο της εισηγήτριας, αλλά και την ανάγκη ε, που έχει τονίσει και η Κομισιόν αλλά και η υπηρεσία μας να υπάρχει μια λεπτομερής νομοθεσία σχετικά με κάποια θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Τώρα, όσον αφορά την ανωνυμία, την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια των δεδομένων, υπάρχει μια ανάγκη να υιοθετήσουμε μια σαφή ξεκάθαρη ε, γραμμή, ένα πλαίσιο ξεκάθαρο, να μιλάμε με, συγκεκριμένες, με συγκεκριμένη γλώσσα, χωρίς κάτι το διφορούμενο. Όπως έχουμε πει και από τη, στο κείμενό μας ε, της 5ης Μαρτίου που δημοσιεύεται και στο website μας, η προστασία των δεδομένων δεν είναι ένα εμπόδιο για να δημιουργήσουμε μία άμεση και αποτελεσματική μεταφορά οργάνων. Ίσα ίσα η προστασία των δεδομένων θα βελτιώσει τις ε, την ποιότητα των πληροφοριών, το, την διαθεσιμότητα των πληροφοριών, την αξιοπιστία των πληροφοριών. Και κάποια από τα σχόλιά μας, σχόλια τα οποία έχω συμπεριλάβει στο κείμενο της 5ης Μαρτίου, ε, συνηγορούν υπέρ μιας αλλαγής της γλώσσας και όχι υπέρ κάποιων ουσιαστικών αλλαγών στο κείμενο, στην πρόταση. Επίσης προτείνουμε να ενισχύσουμε το γενικό επίπεδο ασφάλειας και να συμπεριλάβουμε στην οδηγία κάποιες αναφορές σε συγκεκριμένα μέτρα ασφάλειας να, γίνεται, να γίνει σαφής ανάλυση του κινδύνου και των, της ε, επίσης θα πρέπει να δούμε και το μέλλον. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τα, τις διαφορετικές δυνατότητες, τα διάφορα επίπεδα ε, για να διασφαλίσουμε την ανωνυμία των δεδομένων και των πληροφοριών, κυρίως όσον αφορά την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Χαιρόμαστε που η πρόταση συμπεριλαμβάνει και μία αναφορά στην ανάγκη να συμβουλευόμεθα τις εθνικές αρχές για την προστασία των δεδομένων, κυρίως αναφορά τη μεταφορά των οργάνων σε τρίτες χώρες. Επίσης, ε, γίνεται και άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά στο άρθρο 18.2 ΣΥΓΜΑΤΑΦ. Είναι ένα μήνυμα συνεργασίας ανάμεσα στις εθνικές αρχές είναι ένα σημαντικός κανόνας ε, γιατί όπως μπορείτε να δείτε η προστασία, οι αρχές για την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να δούμε τι, ε, ποιες είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων. Τώρα, κάτι άλλο, Πρόεδρε, αφορά το, την πολιτική για τα δικαιώματα πρόσβασης. Το βασικό σχόλιο που θέλουμε να κάνουμε ε, σχετίζεται με την ιχνηλασιμότητα, με την ανωνυμία. Καταλαβαίνουμε ότι ο στόχος της πρότασης είναι να εξασφαλίσει ένα καλύτερο επίπεδο ιχνηλασιμότητας, αν θέλετε, των ε, πληροφοριών να, ε, ε, ταυτόχρονα όμως να έχουμε και ένα ε, αξιόπιστο σύστημα για, την, για τον εντοπισμό των οργάνων και των δοτών. Η ανωνυμία υπό το φως της οδηγίας 9546 σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε τα δεδομένα, δεν αναγνωρίζουμε τα άτομα. Εδώ όμως μιλάμε για εμπιστευτικότητα Μιλάμε για το απόρριτο που θα αφορά κάποιες πληροφορίες, κυρίως όσον αφορά τον δότη, όχι όμως για πλήρη ανωνυμία. Επομένως θα δείτε ότι στην χωμοδότηση της υπηρεσίας μας ε, υπάρχουν κάποιες προτάσεις ε, που αφορούν κάποια εκτιμώντας και κάποια άρθρα και είμαστε στη διάθεσή σας να κάνουμε οποιασδήποτε άλλες διευκρινήσεις ή τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, εμείς είμαστε εδώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σορνόσα Μαρτίνε, η σκιώδη συγγύτρια τη Σοσιαλιστική Ομάδα, είναι εδώ. Θέλω να σα ζητήσω εάν σα ενδιαφέρει να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μπρεπούλς για το έγγραφο εργασία που μας έχει παρουσιάσει. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία περιλαμβάνει το έγγραφό της. Έχουμε συνεργαστεί και σε άλλες ευκαιρίες για το θέμα αυτό και γνωρίζω ότι έχει συλλέξει πολλές πληροφορίες, τις έχει επεξεργαστεί ενδελεχώς και το κείμενό της μου άρεσε. Νομίζω ότι όλοι μπορούν να συμφωνήσουν σε σχέση με τους στόχους αυτής της οδηγίας δηλαδή να αυξήσουμε τη διαθεσιμότητα οργάνων, να βελτιώσουμε την ασφάλεια των μεταμοσχεύσεων και να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι πιο προσιτό το σύστημα μεταμοσχεύσεων για αυτούς οι οποίοι απαιτούν μεταμοσχεύσεις. Τα μέτρα τα οποία προτείνονται λοιπόν για τη δημιουργία μια σειράς από εθνικών αρχών εποπτικού χαρακτήρα, η εξέλιξη μιας κοινή δέσμης μέτρων για την έγκριση των δωρεών και οι προγράμματα για την δωρεά και την μεταμόσχευση οργάνων, όλα αυτά μας φαίνονται ότι είναι απαραίτητα, όπως επίσης και το να εξασφαλίσουμε ένα σύστημα ίχνη λασιμότητος το οποίο θα προπαρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και να υπάρχουν και οι απαραίτητες συναφείς δομές εποπτείας και επιθεώρησης, γιατί και στον τομέα αυτό θα πρέπει να επιφέρουμε βελτιώσεις και να διατηρήσουμε την ύπαρξη των απαραίτητων αυτών δομών. Μου φαίνεται επίσης πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε την προστασία των δωρητών, να διατηρηθεί η, ανωνυμή, η ανωνυμία τους και να υπάρχει η κατάρτιση μητρών για τα όργανα. Συμφωνώ λοιπόν σχεδόν σε, ουσιαστικά σε όλα τα μέτρα αυτά τα οποία μας προτείνει η κυρία Μπρέπουλς και τα οποία περιλαμβάνεται εξάλλου και στην πρόταση της Κομισιόν που θεωρώ ότι είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε αυτή την πρόταση, αν όχι στην τρέχουσα θητεία σίγουρα στην επόμενη, με την επεξεργασία των προτάσεων της Κομισιόν, αλλά προς το παρόν μπορώ να εκφράσω την, ε, την συμφωνία με την κυρία Μπρέπουλς. Υπάρχουν ορισμένα σημεία στα οποία υπάρχει μια ασάφεια ίσως με τη μετάφραση, γι' αυτό θέτω το ερώτημα. Ξέρουμε ότι στην Ευρώπη βέβαια δεν υπάρχουν κοινά πρότυπα ποιότητος και ασφάλειας των οργάνων προς μεταμόσχευση και υπάρχουν και διαφορές σημαντικές στον αριθμό των μεταμοσχεύσεων μεταξύ μιας χώρας και της άλλης. Επειδή αύριο θα ψηφίσουμε μία οδηγία η οποία ασχολείται με τα θέματα της διαμεθοριακής παροχής υγειονομικής φροντίδας, θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Μπρεπούλς αν συμφωνεί να υπάρξει στην οδηγία αυτή που θα ψηφίσουμε αύριο μια εξαίρεση που να καλύπτει τις μεταμοσχεύσεις οργάνων. Γιατί αυτό, γιατί είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές, είναι τόσο μεγάλες οι διακυμάνσεις σε πρότυπα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα με την οδηγία αυτή, αν συμπεριλάβουμε τα θέματα μεταμοσχεύσεως οργάνων, δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια χωριστή αντιμετώπιση για τις μεταμοσχεύσεις. Θα πρέπει να είναι λοιπόν χωριστή η αντιμετώπιση του Δεν ξέρω αν σύμφωνη η κυρία Μπρέπουλς για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι το μόνο σημείο στο οποίο έχω μια αμφιβολία για την εκθεσή της είναι ακριβώς το θέμα της συμπερίληψης ή όχι των μεταμοσχεύσεων στην οδηγία για τις διαμεθοριακές ε, παροχές ιατρικών φροντίδων. Αυτό θα ήθελα να τη ρωτήσω και μόνο λοιπόν. Ευχαριστώ λέει και ο Ευχαριστώ πολύ. Ο καθηγητής Ανδρέας θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πραγματικά ε, σημαντική εργασία που πραγματοποίησε σε σχέση με την έκθεσή της διότι η κάθε οδηγία έχει κοινού στόχους και εδώ πρόκειται για τη διαθεσιμότητα των οργάνων στην Ευρώπη. Οι πραγματικές μεταμοσχέσεις δεν εξαρτώνται μόνο από την ασφάλεια και την ποιότητα του οργάνου και των κανονισμών που διέπουν αυτή τη δραστηριότητα. Είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να μπορούν να προχωρήσουν σε μεταμοσχεύσεις. Και θυμάμαι ε, μια συγκινητική υπόθεση στη Λετωνία. Ένας νέος αυτοκτόνησε όταν τον ειδοποίησαν ότι η πατική μεταμόσχευση ε, που επρόκειται, στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί ακυρώθηκε διότι δεν είχε τα χρήματα για να καλύψει τη δαπάνη και δεν είχε και χρήματα για να πάει σε άλλο κράτος μέλος και ο νέος αυτός αυτοκτόνησε. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την εισηγήτρια να μου πει το εξή Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιήσαμε κανόνες διεθνών οργανισμών για τις μεταμοσχεύσεις. Ας πούμε το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει ήδη συνάψει μια σχετική σύμβαση ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα βιοφάρμακα το 1997. Εκεί ε, προσθέσαν ένα ε, παράρτημα το οποίο ήταν αφιερωμένο αποκλειστικά στις μεταμοσχεύσεις. Έχω εργαστεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης και θυμάμαι ότι περάσαμε πολύ χρόνο για να συντάξουμε αυτό το παράδειγμα και ζητήσαμε και τη συμβολή ε, εμπειρογνωμόνων από όλα τα κράτη-μέλη. Βήμα-βήμα πήγαμε. Ε, λύσαμε πολλά προβλήματα και τώρα μήπως ξαναεπινοούμε τον τροχό, μήπως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη δουλειά που έχει ήδη γίνει στο Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσκληθεί να υπογράψει και εκείνη αυτή τη σύμβαση και ήδη 9 κράτη-μέλη έχουν υπογράψει. 11 κράτη-μέλη έχουν υπογράψει από τα παλιά. Η Μάλτα δεν έχει υπογράψει ακόμη. Πιστεύω λοιπόν ότι έχει γίνει πολύ σημαντική επιστημονική ανάλυση μες στον χώρο του Συμβουλίου της Ευρώπης και ε, ε, ε, δεν βλέπω να αντανακλάται το αποτέλεσμα του Συμβουλίου της Ευρώπης στο έγγραφο το οποίο χρησιμοποιούμε εμείς. Πρόεδρος. Ευχαριστώ καθηγητά Ντρεύς. Άλλος κανείς που θέλει το λόγο. Δεν βλέπω άλλον ομιλητή. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Μπρέπολς για να κλείσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την κυρία Λεγκόφ από την Κομισιόν τον, και, τον κύριο Μπουταρέλη από το, την, τον Οργανισμό Προστασίας Δεδομένων και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που συνέβαλαν με τα σχολιά τους σε αυτή τη συζήτηση. Όσον αφορά αυτά τα οποία είπε η κυρία Μπρούνκο, θα ήθελα να πω ότι όταν αναφέρθηκε Έλεγα λοιπόν ότι όταν αναφέρθηκε στις προσθήκες στους στόχους της οδηγίας σε σχέση με την απόρριψη ε, μεταμοσχεύσεων πράγματι ζητήσαμε από ειδικούς να εξετάσουν τις μεθόδους που ήδη χρησιμοποιούν ε, γιατροί ειδικοί για να προλάβουν την απόρριψη οργάνων που έχουν ήδη μεταμοσχευθεί. Τώρα, ως προς τα ίδια τα όργανα, πρέπει να σας πω ότι καλύπτονται από τη φαρμακευτική νομοθεσία. Ίσως δεν ε, καταλάβαμε ο ένας τον άλλον, η μία την άλλη μάλλον, και χρειάζεται να το συζητήσουμε λίγο ακόμη. Ε, έχω κάποιες ερωτήσεις για τον κύριο Μπουταρέλη, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Το έγγραφό του αναφέρεται στην αοριστία που υφίσταται μεταξύ ανωνυμίας και χνηλασιμότητας. Δηλαδή είναι δύσκολο να συμβαδίζουν αυτά τα δύο. Ίσως χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω λοιπόν στην έκθεσή μας, διότι η ανωνυμία σαν στόχο έχει να μην είναι γνωστός ο δότης στο λήπτη δεν έχει σχέση με τις αρχές ε, ή όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε να είναι χειλάσιμα τα όργανα, αλλά ίσως πρέπει να ορίσουμε μια διαχωριστική γραμμή ή να επιλέξουμε άλλες έννοια, άλλες έννοιες, άλλες λέξεις. Όταν μιλάμε δηλαδή για ηχνηλασιμότητα εφικτή για τις αρχές. Αλλά η ανωνυμία πρέπει να διατηρείται μεταξύ ε, δότη και λήπτη. Έχω και μια άλλη ερώτηση ακόμη. Ε, μου στείλατε ένα υπόμνημα και στην παράγραφο 21 λέτε, προτείνετε μάλλον, ότι για την ηχνηλασιμότητα πρέπει να έχουμε ένα έμεσο σύστημα ταυτοποίησης σαν λύση, αλλά δεν καταλαβαίνω τι θα πει αυτό το έμεσο σύστημα ταυτοποίησης, ε, ταυτοποίησης μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Ακόμη, στο ίδιο υπόμνημα που μας υποβάλλατε, αναφέρεστε στην ανάγκη να μπορούμε να ταυτοποιήσουμε τον λήπτη και η κυρία Μπρούγκο μόλις μας είπε ότι και η Κομισιόν έχει την άποψη ότι ο καταμερισμός δεν αποτελεί τμήμα των στόχων αυτής της συγκεκριμένη οδηγίας και η τακτοποίηση του λήπτη δεν είναι κάτι που πρέπει να μας αποσχολήσει, νομίζω. Ευχαριστώ κυρία Ζανούσα για την υποστήριξή σας και τις ε, πρόσθετες πληροφορίες που μας δώσατε. Τώρα θα είστε και ένα ζήτημα σε σχέση με την αυριανή μας συζήτηση και την ψηφοφορία για την διασυνοριακή περίθαλψη. Και άλλοι συνάδελφοι έχουν ενδιαφερθεί για αυτό το θέμα και έχουν ζητήσει από τον κύριο Μπόης, τον εισηγητή, να μην περιλάβει τα όργανα και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων σε αυτή την οδηγία. Και έχει καλυφθεί αυτό με μια συμβιβαστική τροπολογία για την ψηφοφορία την αυριανή. Ελπίζω ότι θα το υποστηρίξουμε όλοι μας αυτό. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Αντρέας για την πολύ σημαντική ενημέρωση που μας έκανε και τις πρόσθετες πληροφορίες που μας έδωσε για τα, τις σχετικές ε, μελέτες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εξ όσων γνωρίζω, δεν αναφερόμαστε στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο προήμιο της Κομισιόν. Ε, φαντάζομαι όμως καθώς θα συνεχιστεί η διαδικασία οτιδήποτε τεκμηρίωση υφίστατη η οποία θα είναι χρήσιμη για την εφαρμογή και την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας που εξετάζομαι θα περιληφθεί θα την εξετάσουμε και θα τη συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν για τη συμβολή σας. Και ελπίζω ότι θα συνεχιστεί η συζήτηση σε κάποια μεταγενέστερη ημερομηνία. Ευχαριστώ. Thank you very much. If I understand well... Ωραία. Αν κατάλαβα καλά, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που αφορούν τον κύριο Μπουταρέλη. Και θα μπορούσε να θέλετε να απαντήσετε τώρα. Okay, we have time enough. Okay, Mr. Mr. Έχουμε χρόνο. Κύριε Μπουταρέλα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμμερίζομαι απόλυτα, ε, συμφωνώ με τα σχόλια που έκανε η συγγήτρια. Απόρριτα, μυστικότητα, ε, και εμπιστευτικότητα ανάμεσα στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται ανάμεσα στον δότη και στον ελίπτη πλήρη λασιμότητα των ε, πληροφοριών, ε, τουλάχιστον όσον αφορά τα αρμόδια όργανα και που είναι απαραίτητα για τους ελέγχους. Ίσως γι' αυτό να πρέπει να διαγραφεί ένα από τα άρθρα της πρότασης και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 17 διότι το άρθρο αυτό δυστυχώς μιλάει για το ανώνυμον ε, ανωνυμία και, το, και όπως σας είπα και προηγουμένως τα θέματα αυτά καλύπτονται από την οδηγία 9546 και η οδηγία αυτή καθορίζει, ε, αναφέρεται σε μια διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις πληροφορίες, ε, ανάμεσα σε έναν ε, μη εντοπίσιμο ή εντοπίσιμο δότη και στις πληροφορίες που πρέπει να θεωρηθούν ανώνυμες. Εδώ όμως δεν έχουμε να κάνουμε με ανώνυμες πληροφορίες. Αυτό το που χρειαζόμαστε εδώ είναι να αυξήσουμε και να εναρμονίσουμε τα μέτρα σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε μια πιο αυστηρή ε, εμπιστευτικότητα, ε, μια αυστηρή πολιτική εμπιστευτικότητα, όχι όμως να βάλουμε ένα εμπόδιο στο έργο των αρμοδίων οργάνων όταν πρέπει να έχουν την απαραίτητη πρόσβαση στις πληροφορίες. Και θα πρέπει να διασφαλίσουμε και την υγεία και των δοτών και των λιπτών και καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κανένας άλλος δρόμος να ακολουθήσουμε. Επομένως η, η χνηλασιμότητα είναι κάτι το οποίο είναι αντίθετο με την πλήρη ανωνυμία. Δεν θέλουμε βέβαια να αυξήσουμε εμείς την προστασία στα, όσον αφορά τις, τα, τις πληροφορίες στα δεδομένα. Θέλουμε να υποστηρίξουμε το μήνυμα το οποίο βγαίνει από αυτή την πρόταση. Πλήρη, πλήρης και άμεση ροή πληροφοριών που πρέπει να είναι ασφαλής. Τώρα, για το δεύτερο αίτημα, κύριε Πρόεδρε, το σημείο με το οποίο αναφέρθηκε, αφορά μια, ένα από τα μέτρα κωδικοποίησης που ίσως επιτρέψει στα αρμόδια όργανα να έχουν μια πρόσβαση σε πληροφορίες ένα διαφορετικό βαθμό πρόσβασης με διαφορετικά μέτρα. Με ένα κλειδί, παραδείγματος χάρη, ή με έναν άλλον με ένα άλλο σύστημα κωδικοποίησης. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό επίσης είναι ότι θα υιοθετήσουμε ένα ευρωπαϊκό κωδι... σύστημα κωδικοποίησης και η πλήρης πρόσβαση σε ένα σύστημα που θα επιτρέπει την αναγνώριση ενός ατόμου θα γίνεται παρά μόνο εάν και εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο Γι' αυτό ακριβώς το λόγο προτείναμε να δούμε λίγο και το μέλλον, να δούμε τις νέες τεχνολογίες, όχι μόνο όσον αφορά τις παραβάσεις, αλλά και τα εναλλακτικά συστήματα για την κωδικοποίηση των πληροφοριών και ε, να εξασφαλίσουμε μία άμεση και γρήγορη πρόσβαση πληροφορίες εκεί που αυτό χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το θέμα και ας ανοίξουμε το σημείο 5 που είναι η προφορική ερώτηση 2009 03 σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των θρεπτικών συστατικών και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Αουκέν που εκπροσωπεί την κυρία Χάση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ εκπροσωπώ την Σάτου Χάση, που δεν μπορεί να είναι δυστυχώς παρούσα. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι γιατί δεν έχουμε ακόμα πάρει κάποια πρόταση από την Κομισιόν για την αντιμετώπιση των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων. Θα ήθελα λοιπόν να είχαμε πάρει ήδη από τον Ιανουάριο την πρόταση της Κομισιόν και όχι πρόσφατα όπως φαίνεται να έχει γίνει τώρα. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω το ερώτημα προς την Κομισιόν κατά πόσον στην πρότασή της έχουμε αυτήν την ε, πρόταση από την πλευρά του Προέδρου Μπαρόζο και έχει προταθεί από ένα ηγέτη του ΕΛΚ και όχι ένα ηγέτη του, της Κομισιόν. Αυτό μου φαίνεται πολύ παράξενο. Αυτό άκουσα να λέγεται ότι η αγροτοεπιστητική βιομηχανία περίμενε μια θετική απάντηση από την Κομισιόν και ο κύριος Μπαρόσο είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ε, εξαίρεση για τα βασικά διατροφικά προϊόντα, γάλα, ψωμί, φρούτα, Όλα αυτά τα προϊόντα λοιπόν που είναι καλά για την υγεία. <clears throat> Ανεξάρτητα από το πόση ζάχαρη, λίπος, αλάτι έχουν αυτά τα προϊόντα, εγώ θα ήθελα όμως <clears throat> να το ακούσω εκ του στόματος της ίδιας της Κομισιόν αν πράγματι προβλέπεται μια τέτοια εξαίρεση, αν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο από την πλευρά της Κομισιόν και επίσης υπάρχει το θέμα των ορίων για τα διάφορα προϊόντα. Όλα αυτά είναι φήμες ύπος, ίσως, αλλά μπορούμε να θεωρήσουμε ένα προϊόν που είναι για το πρωινό το οποίο έχει 25% ζάχαρη παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι πλούσιο σε ίνες πραγματικά εφητικές μπορούμε να πούμε ότι είναι καλό για την υγεία. Δεν λέω να τα απαγορεύσουμε αυτά τα προϊόντα Θέλουμε όμως ο καταναλωτής να ξέρει ακριβώς τι περιέχουν αυτά τα προϊόντα. Αυτό ήταν το αντικείμενο της πρότασής μας. Η ελπίδα μας ήταν ότι η Κομισιόν θα ακολουθήσει τη θέση του Κοινοβουλίου και θα δώσει αυτές τις πληροφορίες. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι υπάρχει η πρόθεση να υπάρξει μια σειρά εξαιρέσεων για ορισμένα βασικά προϊόντα. Και δεύτερον, αν αυτή η ρύθμιση θα είναι εξίσου χαλαρή όπως το παρελθόν και θα μπορεί να αποκρύπτει ο παραγωγός από τον καταναλωτή το ότι περιέχουν τα προϊόντα αυτά που αγοράζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είναι ο κ. Ματουράκης. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Και στη συνέχεια θα γίνει ανταλλαγή απόψε. Thank you, uh, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Βουλευτή για τις ερωτήσεις που μου απίφθηνε στις υπηρεσίες της Κομισιόν. Ε, επεξεργαζόμαστε αυτό το θέμα. Από το τότε τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός για τα, τις θρεπτικές ε, αυτό εδώ και κάποιο διάστημα. Πρώτα απ' όλα υπήρχε ένα αίτημα από τον Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον, Ιανουάριο, του 2008. Από τότε η Κομισιόν οργάνωσε πολλές συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη-μέλη. Συζητήσαμε τα ενδεχόμενα, τις ενδεχόμενες για τα θρεπτικά προφίλ λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια τα οποία τίθενται στον κανονισμό. Το ζήτημα λοιπόν αυτό έχει σχολιαστεί εκτενώς, έχουν γίνει παρατηρήσεις από πολλές πλευρές, έχει προκαλέσει πολιτικό ενδιαφέρον στο ανώτατο επίπεδο. Οι συζητήσεις συνεχίζονται στην Κομισιόν και στις υπηρεσίες της Κομισιόν και κατά συνέπεια τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι έτοιμα για να υποβληθούν προς εξέταση στο Ευρωκοινοβούλιο και δεν θα είναι έτοιμα πριν από τις εκλογές του Ιουνίου. Δηλαδή μιλάμε πλέον για το νέο κοινοβούλιο. Η Κομισιόν θα υποβάλει μια πρόταση η οποία θα λάβει υπόψη της το σημαντικό ρόλο ορισμένων τροφίμων και ορισμένων κατηγοριών τροφίμων που αποτελούν βασικά θρεπτικά στοιχεία της διατροφής. Βεβαίω, θέλουμε να έχουμε εξαιρέσεις όπως προβλέπεται και από τον κανονισμό. Τρόφιμα όπως το κρέας, το ψάρι, τα φρούτα, το γάλα, τα αυγά και παραδοσιακά αρτήματα θα εξαιρούνται από την εφαρμογή των προφίλ θρεπτικών ουσιών. Τώρα, όσον αφορά επεξεργασμένα προϊόντα, είτε με βάση το κρέας είτε το τυρί, και εδώ πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό ε, μεταξύ του νοπού κρέατος και των επεξεργασμένων προϊόντων κρέατος, Λοιπόν, τα επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος και τα τυριά θα εξεταστούν ξεχωριστά ώστε να εξασφαλίσουμε παραδοσιακά προϊόντα μέσα από αυτές τις κατηγορίες να συνεχίσουν να έχουν αξιώσεις χωρίς να αμφισβητείται η σύνθεσή τους με την δημιουργία αυτών των θρεπτικών προφίλ. Αυτόν τον τρόπο, κύριε Πρόεδρε, θα ασχοληθούμε με αυτά τα προφίλ περισσότερο σε σχέση με τα επεξεργασμένα προϊόντα που αποτελούν σημαντικό μέρος της διατροφής. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα περισσότερης καινοτομίας και αναδιατύπωσης, αν θέλετε, εκ μέρους της ε, επισητιστικής βιομηχανίας. Η Κομισιόν θεωρεί ότι η αρχή των θρεπτικών προφίλ που συζητήθηκε και περιλαμβάνει περιλαμβάνεται στον κανονισμό που εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι πολύ σημαντικός. Συνεπώς θα προσπαθήσουμε να υποβάλουμε ε, μέτρα σε μορφή σχεδίου ευθυγραμμισμένα με τον κανονισμό και αναλογικά λαμβάνοντας υπόψη το στόχο των μέτρων αυτών και την επιρροή που θα έχουν ε, στις επιχειρήσεις πλέον. Θα ήθελα ακόμη να υπογραμμίσω κύριε Πρόεδρε ότι τα θρεπτικά προφίλ αυτά δεν θα ανακοινώνονται περσέ στους καταναλωτές με αυτή τη μορφή. Η ανακοίνωση προς τους καταναλωτές σε σχέση με τη θρεπτική αξία ορισμένων προϊόντων γίνεται συνήθως μέσω ε, των ενδείξεων πάνω στη συσκευασία και θα έχουμε βεβαίως και προτάσεις για τους καταναλωτές, προτάσεις που το νέο εκλεγέν κοινοβούλιο θα εξετάσει. Εφόσον δεν προλαβαίνουμε για την πρώτη ανάγνωση με αυτό το κοινοβούλιο. Και αυτό είναι σημαντικό που σας λέω, διότι οι καταναλωτές δεν θα έχουν να αντιμετωπίσουν τα θρεπτικά προφίλ με την τυπική τους μορφή. Η ιδέα είναι ορισμένα, τα θρεπτικά αυτά προφίλ να δώσουν τη δυνατότητα σε ορισμένα προϊόντα να γύρουν αξιώσεις. Το, οπωσδήποτε η σήμανση είναι σημαντική στη συσκευασία, αλλά δεν θα δίνουμε πλήρης πληροφορίες όσον αφορά την τρέπτικη αξία των εν λόγω προϊόντων. Όσον αφορά τώρα το θέμα, κύριε Πρόεδρε, της επιστολής που απευθύνθηκε από τον πρόεδρο Μπαρόζο δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω. Γιατί και πώς δηλαδή δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω. Φαντάζομαι ότι είναι αυτονόητο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, δύο ονόματα έχω στο κατάλογο. Κυρία Κόρβε και η κυρία Ροτ Έχετε το λόγο, κυρία Κορή. Κόρη. Whatever. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους προαλήσαντες. Υποστηρίζω πλήρως ε, την ερώτηση και ευχαριστώ και την Κομισιόν για την απάντηση που έδωσε. Θα ήθελα όμως ε, να κάνω και μια περαιτέρω ερώτηση. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε την ΕΦΣΑ η οποία δημιουργήθηκε και η οποία έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και ένας από τους στόχους της ήταν να εξετάσει τα τρόφιμα, την ασφάλεια των τροφίμων ε, που έπρεπε να αντιμετωπιστεί και να εξεταστεί με έναν τρόπο πλήρως αντικειμενικό και όχι μόνο συναισθηματικό ή πολιτικό διότι όλα αυτά τα θέματα, αν θέλετε, ε, απευθύνονται και στο συναισθηματικό και στο μας ε, κόσμο και έγινε και τώρα ούτως ή άλλως υπάρχει στην Πάρμα η υπηρεσία αυτή και θεωρώ ότι τα πράγματα μπορούν να συζητηθούν πολύ πιο αντικειμενικά. Όλο αυτό το συγκινησιακό φορτίο νομίζω σε πολιτικό επίπεδο δεν βοηθάει και ακόμα και ο πρόεδρος Μπορώ Μπαρόζο ασχολήθηκε με τα θέματα αυτά και διαρωτώ με μήπως ακολουθούμε έναν ασφαλμένο δρόμο και μήπως θα τα έπρεπε η ΕΦΣΑ να κάνει όλο αυτό τον, όλη αυτή τη δουλειά. Διότι στο κάτω-κάτω έχουμε δημιουργήσει την υπηρεσία αυτή, ας αφήσουμε να κάνει την δουλειά τους. Γιατί αλλιώς, επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι ακολουθούμε λανθασμένο δρόμο δεν θα καταλήξουν πουθενά. Άκουσα πάρα πολύ προσωπικά την απάντηση και τις εξαιρέσεις ε, που θα δοθούν για τα αυγά, για τα προϊόντα ε, ε, που αφορούν τα ψάρια, τα, τα, το κρέας κτλ. πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε καθαρά τον στόχο μας, τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν αυτά τα προφίλ τα προφίλ αυτά αποφασίστηκαν για να μην δίδονται λανθασμένες πληροφορίες ε, για τα προϊόντα, να μην θεωρούμε ότι κάποια προϊόντα είναι υγιεινά ενώ δεν είναι. Γι' αυτό θεωρούμε ότι όσον αφορά τα αυγά, τα ψάρια, τα προϊόντα με βάση το κρέας, ε, είπατε ότι εξαιρούνται, αποκλείονται. Ε, δηλαδή δεν, θα, δεν υπάρχει θέμα υγείας όσον αφορά όλα αυτά τα προϊόντα. Συμφωνώ Συμφωνείτε με το συμπέρασμα αυτό. Το γάλα και τα αυγά και όλα αυτά τα εξαιρούμενα προϊόντα δεν θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή να, υπάρχει, να υπάρχουν πληροφορίες συγκεκριμένε. Επίσης είπατε ότι τα προφίλ αυτά των τροφίμων δεν παίζουν κανένα ρόλο όσον αφορά την προστασία, ε, ενημέρωση του καταναλωτή. Εγώ θεωρώ ότι είναι κρίμα αυτό, διότι αν έχουν δημιουργήσει αυτά τα προφίλ και εάν υπάρχει και ένας ελάχιστος κοινό παρονομαστής ε, για όλα τα προϊόντα, θα πρέπει να κάνουμε και μία περαιτέρω προσπάθεια να ενημερώσουμε τους καταναλωτές όσον αφορά τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές των τροφίμων. Δηλαδή θα, θα πρέπει να ε, τονίσουμε κάπως αυτό τον, ε, και τον επικοινωνιακό τομέα. Είναι κρίμα που δεν ασχολούμεθα με την με τον επικοινωνικό τομέα και να ενημερώσουμε περισσότερους καταναλωτέ για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Η κυρία Ροτ Μπέρεντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να επανέλθουμε στο θέμα του γιατί καταρχήν προτάθηκε αυτή η νομοθεσία για το θέμα αυτό. Η νομοθεσία έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει τα θέματα της προσθέμενης αξίας. Δεν έχει να κάνει με την ακρίβεια ή όχι των διατυπώσεων που περιλαμβάνονται μέσα στα, στις ετικέτες. Είναι πολύ δύσκολο πραγματικά να αποδείξει κανείς επιστημονικά ότι ένα προϊόν είναι καλό για το κυκλοφοριακό ή για τη χόρεψη ή για οτιδήποτε άλλο ή ότι υπάρχει μια ουσία παγκοσχάρη η οποία μειώνει τον κίνδυνο από την υψηλή χολυστερίνη. Δεν υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να έχουμε απόλυτα επιστημονικά να εδραιώσουμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ. Δεν είναι θέμα επομένως να υπάρχει κάποια ένδειξη σε σχέση με την υγεία ή όχι. Και εγώ συμφώνω με την Κομισιόν Μπορεί να πει κανεί ότι το χαμομήλι έτσι, χαλαρώνει τον ανθρώπινο οργανισμό. Τέτοια γενικά πράγματα μπορεί να πει κανεί, Ναι. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω ιδιαίτερα τη λογική αυτών των προφίλ για την αξία που έχουν τα προϊόντα αυτά, την θρεπτική αξία. Δεν ξέρω λοιπόν με ποιο τρόπο έχουν συνταχθεί και αυτά τα προφίλ για την θρεπτική αξία και έχουμε τον Οργανισμό για την Τροφιμική Ασφάλεια, έχουμε την ΕΦΣΑ, η οποία ασχολείται με τα θέματα αυτά. Αυτό το οποίο έχει πράξει τώρα η ΕΦΣΑ όλα αυτά τα χρόνια καλύπτεται από ένα πυκνό πέπλο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Ο διευθυντής της ΕΦΣΑ, της τροφιμικής, εταιρείας τροφιμικής ασφάλειας, έχει έρθει μας και όταν τον ρωτήσαμε πώς ακριβώς συντάσσεται αυτά τα προφίλ θρεπτικής αξίας, και αυτό πριν από 6 ή 7 χρόνια είχε αναλάβει αυτό το, είχε αναλάβει αυτό το έργο, είπε όταν μας ζητηθεί θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Και ο νέος διευθυντής της ΕΦΣΑ δεν έχει αλλάξει τίποτα σε όλα αυτά. Προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω τι γίνεται. Έχουμε λοιπόν προϊόντα, 200 προϊόντα, τα οποία έχουν όλα ε, ζάχαρη ή πολύ αλάτι, τα κονφλέξ, πούμε, αυτά που τρώμε κάθε μέρα ποιο είναι τελικά το θρεπτικό προφίλ ενός ε, συσκευασμα, μιας συσκευασίας cornflakes. Τι μπορούμε να πετύχουμε τώρα, τι μπορούμε να συναγάγουμε από αυτά τα οποία υπάρχουν σε τεχνικό επίπεδο, σε επιστημονικό επίπεδο, τι μπορούμε να βγάλουμε από αυτά τα στοιχεία. Εγώ συμφωνώ σε πολλά σημεία με τον κύριο Μαθιουδάκη. Νομίζω και οι δύο έχουμε παρακολουθήσει από κοινού αυτό το θέμα στην προσπάθεια να προχωρήσουμε για την νομοθεσία των θεμάτων αυτών. Αλλά είναι κακό κατά την άποψή μου να υπάρχει νομοθεσία σε σχέση με τους ισχυρισμούς που περιέχονται στη συσκευασία των προϊόντων. Το και χρειάστηκε να ε, εξηγήσει η ίδια η Κομισιόν αν, γιατί υπήρχαν ανακρίβειες για τα θέματα αυτά που πρέπει να αντιμετωπιστούν από την ε, νομοθεσία αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει μια προσπάθεια από την πλευρά της Κομισιόν να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά και να έχει μια σωστή διαδικασία επιτροπολογίας. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο προτείνει ο κύριος Μαθιουδάκης είναι σωστό, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Γιατί στην αρχή βάλαν τις φωνές λέγοντας η παραγωγή ελαιολάδου, παραγωγή Εμείς Έχουμε λιπαρά. Τι λιπαρά έχουμε, δεν έχουμε λιπαρά. Μετά η παραγωγή ελαίου, ελαίων από το, του λινελαίου παραγωγή χάρη. Υπάρχει και αυτή. Έχουμε τελείω υγιεινά προϊόντα. Και είπαν άλλοι ότι αυτό δεν είναι θέμα που αφορά τα βασικά προϊόντα, αφορά μονάχα τα συσκευασμένα προϊόντα. Μα με τον τρόπο αυτό δεν μπορούμε να έχουμε μια πραγματική υγειονομική νομοθεσία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει σωστά ο κ. ότι υπάρχουν κάποιες Εξαιρέσει οι οποίες δεν περιλαμβάνονται εδώ στην ε, νομοθεσία. Και σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμού που περιέχονται στη συσκευασία και στην, ε, στο προφίλ το υγειονομικό, το θρεπτικό μάλλον προφίλ αυτών των ουσιών, εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει κάποια αντιστοιχεία μεταξύ αυτών που αναφέρονται στη συσκευασία και των προϊόντων, των ιδιωτήτων των προϊόντων αυτών. Εμείς θεωρούμε ότι αν το θρεπτικό προφίλ πράγματι δεν πραγματοποιείται από το προϊόν αυτό, θα πρέπει να υπάρχει κάποια προειδοποίηση στην συσκευασία για τα θέματα αυτά. Και έχουμε εδώ μία σειρά εξαιρέσεων, μερικών εξαιρέσεων από την ε, ρύθμιση αυτή. Εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση για τα επεξεργασμένα ε, προϊόντα. Και από αυτά τα οποία είπε ο εκπρόσωπος της ΕΦΣΑ δεν έχω καταλάβει. Άμα τα αντιμετωπίζετε αυτά τα προϊόντα, τι κάνετε. Κατατίζετε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, όλα τα γιαούρτια μαζί, όλα τα έλαια μαζί. Πώς μπορείτε εσείς να αποφασίσετε ποιο είναι ένα καλό θρεπτικό προφίλ έχει να κάνει με το ίδιο το προϊόν, έχει να κάνει με την άποψη των επιστημόνων που λένε πόσο παραγωγικά λιπάρα πρέπει να έχει ένα γιαούρτι ή όχι. Ποια, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε. Εγώ θα ήθελα να ξέρω. Για μένα μπορεί να είναι 1% λιπαρά, ο άντρα μου μπορεί να θέλει 3,5% λιπάρα στο, στο γιαούρτι. Που λέει ότι αυτό είναι καλύτερο. Εσεί πώ θα το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα. Να δούμε έναν τρόπο λοιπόν με τον οποίο θα μπορέσουμε με λογικό τρόπο να έχουμε κάποιες προσδοκίες σε σχέση με τη δημιουργία αυτών θρεπτικών Thank you very much. Ευχαριστώ. πολύ. Ο κύριος Σόκερ και πάλι. Η κυρία Σόκερ, με συγχωρείτε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την απάντηση που μου έδωσε η οποία κάπως αν θέλετε επιβεβαίωνει ουσιαστικά τις φήμες που έχω ακούσει δηλαδή σωστά άκουσα ότι αυτό το οποίο μας φημί λέγεται ότι συνέβη, έχει πράγματι συμβεί. Ακούγοντας και την Τάκμαν τώρα, πρέπει να σας πω ότι τελικά μας αφήνουν πολύ λίγο χρόνο. Είναι τα πράγματα τόσο περίπλοκα, είναι τόσο δύσκολο να έχει κανείς ενημέρωση όσον αφορά αυτά τα θρεπτικά προφίλ θα μπορούσαμε να είχαμε κάποια σαφή απάντηση ώστε να γνωρίζουμε ότι ε, πάνω στο τάδε προϊόν δεν μπορεί να υπάρχει ο ισχυρισμός ότι είναι καλό για την υγεία εφόσον υπάρχουν συστατικά τα οποία το καθιστούν ακατάλληλο για την υγεία. Ένα προϊόν είναι καλό γιατί έχει πάρα πολλέ ίνες, αλλά αν έχει και πάρα πολύ ζάχαρη, τι γίνεται. Είναι καλό για την υγεία. Λοιπόν, ουσιαστικά νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε πρώτα απ' όλα να δούμε τι θα μας στείλει η Κομισιό. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να επισημάνω ότι παρακολουθούμε πολύ στενά τα δραματιζόμενα, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό οι καταναλωτές να έχουν αξιόπιστες πληροφορίες όσον αφορά τα περιεχόμενα ε, των τροφίμων τους. Δεν πρέπει δηλαδή να υπάρχουν αξιώσεις ή ισχυρισμοί που να τους οδηγούν σε λάθος επιλογές. Θα ζητήσουμε λοιπόν από την Κομισιό η ανακοίνωση να τηρήσει κανόνες πολιτικής ουδετερότητας όταν, ε, δηλαδή και να μην απευθύνεται σε ένα κόμμα αλλά να απευθύνεται στην αρμόδια επιτροπή η ανακοίνωση της Κομισιό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, τώρα ο κύριος Χασίμπα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με πολλούς από αυτούς που έλαβαν το λόγο ότι είναι σημαντικό ο πληθυσμός να έχει θρεπτικά προϊόντα και υγιεινά προϊόντα. Αυτό δεν, δεν νομίζω ότι κανείς το διαφυσβητεί. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της ε, παχυσαρκίας στον πληθυσμό. Πρέπει να δώσουμε την πρέπουσα προσοχή σε αυτό το θέμα και την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι ο κατάλληλος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε είναι με τα προφίλ θρεπτικής αξίας και με τους ισχυρισμούς που βρίσκονται πολλές φορές στα προϊόντα. Και όπως και η κυρία Ροτμπέρεν θα, ήξερα εγώ, θα ήθελα εγώ να ξέρω βάσει ποιων επιστημονικών εμπειρογνωμών συνών μπορεί η Κομισιόν να προχωρήσει στη διατύπωση αυτών τον προφίλ. Νομίζω ότι πολύ λίγα πράγματα από αυτά που λένε οι επιστήμονες είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ξέρουμε ότι είναι θετικό. Παραδείγματος χάρη ότι τα φρούτα και τα λαχανικά είναι θετικά και ότι προστατεύουν σε κάποιο βαθμό από τον καρκίνο. Αλλά είναι λίγα τα πράγματα τα οποία είναι πραγματικά εδρεωμένα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Κομισιόν να ξέρω πώς αιτιολογεί όλα αυτά τα προφίλ τα οποία δημιουργεί αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι μονάχα τα προϊόντα τα οποία, τα συγκεκριμένα τα οποία ε, τρώγονται, μέσα από τον καταναλωτή αλλά το συνολικό πλέγμα όλων αυτών των προϊόντων τα οποία αλληλεοεπιδρούν μεταξύ τους μέσα σε ένα διατροφικό σύστημα. Νομίζω ότι η καθημερινή ζωή μας δείχνει ότι υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές στο διατροφικό τομέα. Θα ήθελα να ξέρω και αν η Κομισιόν έχει προχωρήσει περισσότερο από το διατροφική μελέτη, αν έχει κάνει μελέτες ψυχολογικού χαρακτήρα, πώς τελικά, παραγματικά, αυτά τα οποία λέγονται οι παροιμίες, οι παραδόσεις οι οποίες υπάρχουν για, τη διατροφική, και τις διατροφικές συνήθειες αν έχουν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα και πολλές φορές αντικρούν τις ε, επιστημονικές εμπειρογνωμοσύνες. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να έχουμε μια παράδοση σε σχέση με τη χρήση των τροφίμων η οποία βασίζεται στην παράδοση και στις εθνικές συνήθειες. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν πώς αντιμετωπίζει αυτό το φαινόμενο η Κομισιόν και ιδίως όταν υπάρχουν συγκρούσεις με αυτό το οποίο μπορεί κανείς να συνάγει από τη διατροφική αξία οτιδήποτε άλλο. Ποια είναι λοιπόν η... με, ποιο τρόπο προσπαθεί η Κομισιόν να ζυγίσει αυτές τις διαφορετικές απόψεις και να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Thank you very much. Πρόεδρο, σε ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρενάτα Ζούμα είναι η τελευταία ομιλήτρια στον κατάλογο μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ ζητώ συγγνώμη γιατί άργησα, ήμουν μπλοκαρισμένο στον αυτοκινητόδρομο. Κρίμα που δεν ήμουν παρούσα να ακούσω αυτά που είπε ο κύριος ε, Μαθιουδάκης. Εγώ θεωρώ όμως ότι αυτά τα οποία λέει η κυρία Ροτπέρεντ ήταν ε, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και ο Ζέμπερ επίσης. Τι είναι τώρα υγιές. Όταν συζητούσαν για πρώτη φορά τους ισχυρισμούς περί υγιεινών προϊόντων, μας είπε η Κομισιόν ότι υπάρχουν φρούτα τα οποία είναι γλυκά, έχουν πολύ ζάχαρη. Αυτό δεν σημαίνει επομένως ότι μπορούμε να εξισώσουμε οτιδήποτε είναι φρούτο με την ε, υγιεινή διατροφή. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα φρούτα τα οποία έχουν πάρα πολύ ζάχαρη και μπορούν μελλοντικά να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα μετά από πολύ μεγάλη κατανάλωση. Επομένω είναι πολύ δύσκολο να έχουμε σαρωτικέ δηλώσει αυτού του είδου στα φρούτα. Είναι υγιή τέρμα. Υπήρξαν λοιπόν πολλέ απόψει που έχουν διατυπωθεί, παραδείγματο χάρη, οι πράσινοι, κάποιοι πράσινοι που λέγανε κάθε μέρα πρέπει να τρώει κανεί χι φρούτα και αυτό είναι ε, καλύτερο ή ότι τα προϊόντα τα οποία έχουν ε, περισσότερα υγρά είναι πιο υγιεινά ή δεν είναι υγιεινά. Λοιπόν, όλα αυτά μας οδηγούν πάρα πολλές φορές σε λαθασμένους δρόμους. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι ανοησίες και μόνο ανοησίες. Χαίρομαι τώρα για το γεγονός ότι τώρα προβλέπονται κάποιες εξαιρέσεις από το γενικό κανόνα όταν εμείς προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τη θρεπτική αξία ορισμένων προϊόντων σε σχέση με τις, οριακές, με τις τιμές κατοφλίου για το αλάτι και τη ζάχαρη. Νομίζω ότι αυτά τα προϊόντα ε, θρεπτικής ε, αξίας θα πρέπει να βασίζονται στα, θα πρέπει να αφορούν κυρίως τα βασικά προϊόντα. Κύριε Μαθιουδάκη, είχαμε ήδη ασχοληθεί εδώ και τρία χρόνια με το θέμα του ψωμιού. Έχουμε πει ότι το ε, λευκό ψωμί χάρη που καταναλώνεται στην Νότια Ευρώπη δεν μπορεί να εξισωθεί με το μαύρο ψωμί το οποίο τρώμε πολύ περισσότερο στη Βόρεια Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε λοιπόν τι ακριβώς είναι υγιεινό και τι όχι, γιατί είναι τόσο μεγάλη η πολυμορφία της διατροφής και του τρόπου ζωής στην Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολλές περιφερειακές και τοπικές σπεσιαλιτέ και αυτό είναι κομμάτι της κουλτούρας μας, ότι υπάρχουν αυτές τις περιφερειακές συνταγές ή τα περιφερειακά προϊόντα, τα οποία επί χιλιάδες χρόνια τα έχουμε στο τραπέζι μας και δεν μας έχουν οδηγήσει ορισμένε από εμά στο θάνατο νωρίτερα. Επομένως, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και πάλι ότι δεν μπορούμε με μια ετικετοποίηση και μια κατάταξη των τροφίμων να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υγεία που μπορεί να προέρχονται από τη διατροφή. Όπω παραδείγματο χάρη υπάρχει Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μονάχα με στατίες διαφώτιση και δεν έχει νόημα λοιπόν να αντιμετωπίσουμε μονάχα τα τρόφιμα αυτά τα οποία παίρνει ο καταναλωτής πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τον τρόπο παραγωγής από τη, από τη γεωργία. Επίσης οι ισχυρισμοί για υγιεινότητα, για υγιειν, η διατροφή των προϊόντων όπως των συγκομισιών θα πρέπει να είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουν ότι δεν παραπλανούν τον καταναλωτή και αυτό είναι θέμα διαφήμιση της διαφήμισης που συνοδεύει αυτά τα προϊόντα. Ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε μία υγιεινή και θρεπτική διατροφή, προϊόντα τα οποία έχουν θρεπτικό χαρακτήρα. Επομένως δεν έχει νόημα να λέμε ότι κάποια προϊόντα είναι αρνητικά και δεν είναι καλά για τον καταναλωτή. Η, η αγορά είναι αυτή η οποία αποφασίζει η ζήτηση των καταναλωτών. Δεν είναι η πολιτική απόφαση η οποία θα μπορέσει να πει αυτό είναι υγιεινό, αυτό δεν είναι. Και εξάλλου δεν υπάρχει επιστημονική βάση όπως έχουμε πει. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι ένα ένα προϊόν είναι θετικό, ένα άλλο όχι. Γιατί έχουμε μια συνολική διατροφή όπου πρέπει όλα τα προϊόντα αυτά να συμμετέχουν και δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τη σημασία των τροφίμων χωρίς να ξέρουμε το συνολικό στυλ ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό οδηγεί σε πλάνες πολλές φορές η δημιουργία των θρεπτικών προφίλ και στην περίπτωση λοιπόν των ε, βασικών προϊόντων, στην περίπτωση των, ε, περιφερειακών και τοπικών σπεσιαλιτέ, βλέπουμε ότι αυτό δεν μπορεί να ακολουθηθεί. Και επίσης δεν μπορούμε να περιμένουμε από την εταιρεία για την ασφάλεια, από τον φορέα για την ασφάλεια των τροφίμων, για την ΕΦΣΑ, από μόνη της να αποφασίζει μονομερός για τις οριακές τιμές, τιμές κατοφλίου, για ζάχαρη ή για, άλλα, για, για Δεν μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο θέμα το οποίο είναι περισσότερο πολιτικού χαρακτήρα σαν να είναι ένα θέμα στο οποίο υπάρχει μια εδρεωμένη επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη. Δεν νομίζω ότι είναι αρνητικά τα τρόφιμα, ότι είναι βλαβερά τα τρόφιμα τα οποία έχουμε στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι είναι καλή η νομοθεσία που ισχύει για τα τροφιμικά θέματα στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποια από τα τρόφιμα τα οποία βρίσκονται στην ευρωπαϊκή αγορά για βλαβερά. Εγώ επομένως θα ήθελα να εξασφαλίσουμε ότι μέσα στη συνολική αυτή είναι του θρεπτικού προφίλ των τροφίμων να υπάρξει και η δυνατότητα εξαιρέσεων ώστε ο καταναλωτής να μην έχει μια αντική εικόνα για το ρόλο της Ευρώπης. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε και στην επόμενη θητεία να εξετάσουμε τη νέα οδηγία για την ε, ετικετοθεσία και την τακτοποίηση των τροφίμων να δώσουμε και μια μεγαλύτερη βάση επιστημονική σε, στις διατυπώσεις που έχουμε και κυρίως τα θρεπτικά προφίλ τα οποία δεν έχουν καμία επιστημονική βάση να μην προωθούνται με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Άουκεν. Α, η κυρία Άουκεν θέλει το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Δεν θα ξανανοίξουμε τη συζήτηση ολόκληρη, εγκρίναμε ό,τι εγκρίναμε. Και πρέπει να μείνουμε στην τοποθέτησή μας. Το να πούμε τώρα, τα φρούτα είναι καλά για την υγεία. Έχουμε μια μεγάλη ομάδα ατόμων που υποφέρουν από διαβήτη τύπου 2. Λοιπόν, αυτοί θεωρούνται άνθρωποι που έχουν καλή υγεία, αλλά παρόλα αυτά τους προειδοποιούν οι ιατροί να μην χρησιμοποιούν, να μην καταναλώνουν μάλλον ορισμένα φρούτα. Τα πορτοκάλια έχουν λιγότερο ζάχαρη από άλλα φρούτα. Λοιπόν, υπάρχουν γενικές ενδείξεις που μπορούν να δοθούν ώστε οι άνθρωποι να μην πεθαίνουν. Πρέπει να έχουν έναν τρόπο τέλο πάντων να γνωρίζουν τι περιέχει ένα προϊόν. Αυτό είναι ο στόχος. Το να λέμε ότι είναι κάτι πρωτότυπο άρα ή παραδοσιακό άρα είναι καλό για την υγεία αυτό δεν ισχύει. Πρέπει να υπάρχουν πληροφορίε και όχι ισχυρισμοί. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπε η κυρία Κόρμπετ. Αν υπάρχουν εξαιρεσει. Οι εξαιρέσει θα πρέπει να αφορούν τους ισχυρισμούς ότι κάτι είναι υγιεινό. Εάν η περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι υψηλή, αυτοί που έχουν χωριστερόλοι δεν πρέπει ε, να καταναλώσουν αυτό το προϊόν. Αλλά πώς θα το γνωρίζουν. Ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει ε, τη ζωή που θέλει βέβαια, αλλά τουλάχιστον να επιλέγει πεφωτισμένα. Πολύ ωραία. Έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα μπορούμε να το ζητήσουμε όλο το θέμα σε όλες τις, ε, με όλες τις λεπτομέρειες και αν κάποιος ε, έχει βαρεθεί με τα φρούτα, δεν να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά και αυτό μπορεί να συμβεί. Κυρία Ζόμερ, πάρα πολύ σύντομα να δώσω μια απάντηση. Τα συστατικά των τροφίμων. Αυτό καλύπτεται από την οδηγία για την ετικετοθεσία. Τι περιέχουμε τα τρόφιμα. Πάντα το έχουμε υποστηρίξει αυτό. Αλλά άλλο το να λέμε τι περιέχεται σε, στα τρόφιμα και άλλο η αξιολόγηση της θρεπτικής ή όχι αξίας αυτών των προϊόντων. Εμείς κάνουμε νομοθεσία για τον μέσο ε, καταναλωτή. Ο μέσος καταναλωτής έχει μία μέση υγεία. Δεν μπορούμε εμείς να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες όλων των ομάδων ασθενών οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα, πραγματικά το διαβίδι που αναφέρθηκε και οι οποίοι χρειάζονται μια ειδική ετικετοθεσία. Δεν είναι δυνατόν. Εμείς αντιμετωπίζουμε μόνο τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε μια μέση κατάσταση υγείας. Αυτό μόνο μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να καλύψουμε όλους τους ασθενείς ή όλους τους ανθρώπους. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν διότι έχουν ειδηθεί τόσο πολλές ερωτήσεις που πρέπει να είστε πολύ απασχολημένος να σημειώνετε κύριε Μαθιουδάκη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν τολμώ να φανταστώ τι ερωτήσεις θα πέσουν όταν θα έχουμε ένα σχέδιο κειμένου μέτρων στο Κοινοβούλιο. Εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα των μελών. Κυρία Κόρμπη, πρώτον πρέπει να αποσαφηνίσω ότι όταν μιλάμε για τις εξαιρεσει, όπως προβλέπετε στον κανονισμό, εννοούμε εξαιρεσει από την ανάγκη να υπόκειται ένα προϊόν στην κατάρτιση ενός θρεπτικού προφίλ. Τα τρόφιμα αυτά λοιπόν τα οποία την χάνουν εξαίρεση δεν είναι υποχρεωμένα να περιλαμβάνουν ένα προφίλ θρεπτικών ιδιωτήτων και θα, επομένως θα υπάρχει δυνατότητα να γίνονται ισχυρισμοί για την αξία τους χωρίς να υπάρχει ο παραμικρός περιορισμός. Αυτό σημαίνει εξαίρεση. Τώρα η απαγόρευση ισχυρισμών περί θρεπτικής ή άλλης αξίας, αυτό βρίσκεται ήδη μέσα στον κανονισμό. Και αυτό αφορά τις, τους ισχυρισμούς όλους τους ισχυρισμούς ε, για τα αλκοολικά ποτά, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορούν να λένε τα αλκοολικά ποτά ότι είναι θετικά, εκτός μονάχα αν αφορούν το γεγονός ότι έχουν μειωμένο ποσοστό αλκοόλ, μειωμένη περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Τώρα εγώ δεν γνωρίζω από εδώ και πέρα τι, θέλετε εσείς. Λέτε ότι πρέπει να υπάρχει και μία επικοινωνία με τον καταναλωτή μέσω των ε, προφίλ θρεπτικής αξίας. Αλλά η κυρία Ζόμερ έδωσε μια απάντηση σε αυτό που είπε στο ερώτημα της κυρίας Άουκεν. Και εγώ τόνισα ότι τα προφίλ θρεπτικής αξίας δεν θα ανακοινώνονται στον καταναλωτή θα είναι μονάχα ένα φίλτρο μέσα από το οποίο μπορεί κανείς να εξετάσει κατά πόσον οι ισχυρισμοί που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα ευσταθούν ή όχι. Και θέλω εδώ να δώσω και μία απάντηση στο ερώτημα του κυρίου Σέμπα. Γνωρίζουμε ότι οι καταναλωτές βασίζουν τις αγοραστικές τους επιλογές σε, σε μια πλειάδα κριτηρίων όχι μόνο η τιμή αλλά και η γεύση, η αισθητική εμφάνιση κτλ. Αλλά όπως συζητήσαμε και όταν εγκρίναμε τον κανονισμό για τα θέματα αυτά, όλο και περισσότερο ο καταναλωτής λαμβάνει υπόψη την θρεπτική αξία, τη διατροφική αξία των προϊόντων. Υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά την σχέση μεταξύ δίαιτας και διατροφής και υγείας και συμφωνώ πάρα πολύ με την κυρία Ζώμεν, αλλά διαφωνώ σε ορισμένα σημεία. Εγώ θεωρώ ότι η παιδεία είναι πρωταρχικής σημασίας. Η πληροφόρηση για τους κατανοτές είναι πρωταρχικής σημασίας. Δεν συμφωνώ λοιπόν ότι, μαζί με την κυρία Ζόμερ ότι η ετικετοποίηση, οι ετικέτες δεν είναι ένας τρόπος πληροφόρησης των καταναλωτών ώστε να μπορέσουν να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές. Νομίζω ότι το αποδέχεται η κυρία Ζόμερ ότι η σωστή περιγραφή στις ετικέτες των προϊόντων θα βοηθήσει πάρα πολύ τους καταναλωτές. Τα θέματα τώρα των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στις ετικέτες, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υποχρεωτικό, έχει ένα εθελοντικό χαρακτήρα και γι' αυτό υπησερχόμαστε με, τις, ε, με τα προφίλ αυτά θρεπτικής αξίας, γιατί κύριε Ζέμπερ, γιατί είναι γεγονός ότι οι ισχυρισμοί που περιέχονται στις ετικέτες επηρεάζουν τους καταναλωτές της επιλογής τους, επομένως ο στόχος των προφίλ θρεπτικής αξίας είναι να εξασφαλίσουμε ότι ο καταναλωτής δεν παραπλανάται με ισχυρισμούς οι οποίοι παρουσιάζουν μόνο τις θετικές πτυχές ενός προϊόντος, ενώ το προϊόν αυτό μπορεί να περιλαμβάνει και αρνητικά στοιχεία. Συμφωνώ βεβαίω μαζί σας και με την κυρία Σόμερ ότι η γενική διατροφή είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τώρα, το τελικό η τελική παρατήρηση. Δεν είναι η ΕΦΣΑ που μπορεί να θέσει τα προφίλ ε, θρεπτικότητας. Θα προσδιοριστούν αυτά από την Κομισιόν. Έτσι λέγεται άλλωστε και στον κανονισμό. Ε, όχι με οποιοδήποτε μορφή επιλέξει η Κομισιόν, κυρία Μπέρ. Υπάρχει περιγραφή σχετική στον κανονισμό. Ε, πρόκειται για επιτροπολογία με εξέταση. Η ΕΦΣΑ βεβαίω θα γνωμοδοτήσει, αλλά στη συνέχεια οι ρυθμιστές που είναι η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη δηλαδή και μετά από εξέταση από το Ευρωκοινοβούλιο θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Νομίζω ότι τα είπα όλα. Α, κάτι ακόμη. Δεν πρόκειται να ε, γίνουν τα προφίλ για εξατομικευμένα προϊόντα. Ε, ο προσανατολισμός μας είναι να έχουμε προφίλ τα οποία να ισχύουν για όλα τα προϊόντα με ορισμένες κατηγορίες τροφίμων που είναι σημαντικές για την γενική διατροφή. Δηλαδή, θα εξετάσουμε ε, το ειδικό πλεονέκτημα κάποιων προφίλ που διαφέρουν από τα γενικά τρόφιμα και που ε, προσφέρουν κάποιο σημαντικό πλεονέκτημα. Okay. Πολύ ωραία λέει ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο-τρία ονόματα ακόμη στο κατάλογο των ομιλητών. Ο κύριος Ζήμπερα. Θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να επαναλάβω το ερώτημα, γιατί δεν έχει απαντήσει η Κομισιόν. Θεωρεί ότι όλοι οι καταναλωτές αποφασίσουν επί τη βάση της λογικής. Έχει κάνει όμως η Κομισιόν μελέτες που να δείχνουν επί τη βάση ποιων κριτηρίων πραγματικά αποφασίζουν οι καταναλωτές. Μπορεί λοιπόν ο εκπρόσωπος της Κομισιόν να λέει ότι είναι ορθολογική η επιλογή των καταναλωτών, αλλά υπάρχουν και μελέτες που καταδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο, ότι δεν είναι ορθολογική. Ποιες μελέτες λοιπόν έχει λάβει υπόψη η Κομισιόν σε αυτήν την περίπτωση. Κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν πρόκειται να ζητήσουμε από την Κομισιό να κάνουν αυτές τις μελέτες. Ε, νομίζω ότι ήδη έχουν πολύ δουλειά στην Κομισιό. Αυτό όμως το που με λυπεί είναι ότι μετά από εντατικό λόμπινγκ φτάσαμε εδώ. Αυτό με ανησυχεί. Δηλαδή μετά από όσα ακούσαμε είναι προφανές ότι ασκήθηκαν τέτοιε πιέσεις ώστε όλα αναβλήθηκαν, αναβλήθηκαν, αναβλήθηκαν και τώρα πάμε για την επόμενη θητεία. Δεν θα πω τίποτα άλλο και ευχαριστώ και την Κομισιόν και αναμένω την απάντηση. Ωραία. Λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μαθιουδάκης, θέλετε να προσθέσετε κάτι σχετικά με την ερώτηση του κύριου Ζήμπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η Κομισιό δεν έχει ζητήσει κάποια συγκεκριμένη μελέτη σχετικά με τη συμπεριφορά των ε, καταναλωτών. Υπάρχουν μελέτες τις οποίες έχει λάβει υπόψη της η Κομισιό. Ξέρουμε ότι τα, όσον αφορά τα, σχετικά με την διατροφή, τα διατροφικά στοιχεία μπορεί να μην ενδιαφέρουν όλους τους καταναλωτές, για κάποιους καταναλωτές όμως είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Αυτό ήταν το τελευταίο σημείο της ε, σημερινής μας ημερήσιας διάταξης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταλλαγή απόψεων και ελπίζω ότι όλοι σας θα είστε παρόντες αύριο, διότι είναι αρκετά φορτωμένο το πρόγραμμά μας. Είναι τελευταία μας συνεδρίαση. Επαναλαμβάνω ότι σας καλώ για την κοινή φωτογραφία κατά διάρκεια του διαλύματος, μεσημεριανού διαλύματος και μετά για ένα ποτό το βράδυ. Ευχαριστώ.